ενημερώσω ότι την Τετάρτη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω τέσσερι πράξεις οι οποίες εγκρίθηκαν στη διάρκεια της συνήθου νομοθετική διαδικασία βάσει του άρθρου 78 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Οι τίτλοι θα δημοσιευτούν